Okay. Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι, μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας. Έχω δίπλα μου την κυρία Κώστα, η οποία θα προεδρεύσει σε ένα μέρο τη συνεδρίασης και περιμένουμε να έρθουν μόνος και οι υπόλοιποι βουλευτέ, αλλά δεν έρθονται. Είναι 9 και 10 και φτάνει πια. Δεν περιμένω άλλο. Καλημέρα σα, καλώ ήρθατε στην κοινή μα συνεδρίαση. Είναι μια μεγάλη χαρά να μπορέσω να προεδρεύσω αυτή τη τελευταία κοινή συνεδρίαση μαζί με την κυρία Κώστα για τα θέματα παιδείας, πολιτισμού και τα λοιπά. Καλώς ήλθατε συνάδελφοι από την Επιτροπή Πολιτισμού και ήτρε, εν πάση περιπτώσει. Πρωτού προχωρήσουμε τώρα στην ψηφοφορία, ας εγκρίνουμε την ημέρα διάταξη. Εάν είμαστε με δίχως παρατήρησης μπορούμε να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Έχουμε λοιπόν την κοινή συνεδρίαση για μια ώρα περίπου. Δεν βλέπω να υπάρχουν παρατηρήσεις. Οι ανακοινώσει μου είναι πάρα πολύ σύντομες. Η συνεδρίαση αυτή μεταδίδεται στο διαδίκτυο και έχουμε σχεδόν όλες τις γλώσσες εκτός από τέσσερις γλώσσες. Λείπαμε γι' αυτό δεν έχουμε ε, σλοβενικά, μαλτέζικα, κροατικά και Εγώ Εδελικά. Και τώρα περνάμε στο σημείο που μας ενδιαφέρει η ψηφοφορία. Η κυρία Κώστα θα αρχίσει την ψηφοφορία μετά από, μέχρι την τροπολογία 2008. Και εγώ θα ξεκινήσω από τη συμβαστική τροπολογία 21. Θα κάνουμε ότι είναι ανθρωπίνως δυνατό, ώστε να προχωρήσει καλά και γρήγορα η ψηφοφορία. Δεν υπάρχουν άλλα σχόλια, κυρία Κώστα. Ευχαριστώ, κύριε Μπούζεκ. Είναι χαρά για μένα να προεδρεύω μαζί σας αυτή την τελευταία κοινή επιτροπή ε, της ΙΤΡΕ και της Επιτροπής Πολιτισμούς για να στηρίξουμε αυτή την πολύ σημαντική έκθεση για, την, ε, τον πολιτισμό και την τομέα τη βιομηχανία. Καλωσορίζω όλου τους ε, συναδέλφους από την Επιτροπή ΚΟΛΤ και ΙΤΡΕ και κυρίως τους δύο συνεισηγητέ, Χέλερ και Μόργαν. Ε, κάναμε μαζί μια έξοχη δουλειά. Εγώ θα πρότεινα στην αρχή να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία και ελπίζω όλοι να έχετε φέρει τις κάρτες σας. Θα πάμε λοιπόν σε μια δοκιμή, μια δοκιμαστική ψηφοφορία. Ξεκινάει η δοκιμή λοιπόν. Δοκιμή, δοκιμή. Πέρας. Εντάξει, εντάξει είμαστε. Ωραία. Ας προχωρήσουμε λοιπόν στη ψηφοφορία μας. Ξεκινάμε λοιπόν. Συμβιβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 113 στην επόμενη σελίδα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 127 στην επόμενη σελίδα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 142, τροπολογία 142 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 143 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 165 στην επόμενη σελίδα. Μίκελς υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 166 ξεχωριστά τμήματα που ζήτησε το ΕΛΚ και οι σοσιαλιστές. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 168 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 12 στην επόμενη σελίδα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 239. Ζητώ συγγνώμη. Α, εντάξει. Πήδηξα μια σελίδα, συγγνώμη. 239 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 190 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 192 κατά τμήματα που ζήτησε το ECR, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 194 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 195 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 218 Μίλναρ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 219 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 221 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές συμβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 232 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 233 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 234 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 14α 14α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 243 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 247 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 248 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 279. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 280. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Και τώρα δίνω το λόγο στον πρόεδρο, στον συμπρόεδρο. Ευχαριστώ κυρία πρόεδρε. Ευχαριστώ Σιλβία. Μπορούμε να συνεχίσουμε λοιπόν. Συμβαστική 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 290 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 297 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 306 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 307 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 308 υπέρ κατά αποχές Απολύπτεται. Συμβαστική 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 317 <clears throat> υπέρ κατά αποχές ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά. 317 ηλεκτρονικά. Πέρα της φοφορίας. Θα δούμε, θα δούμε, λέει ο 318 υπέρ. Κατά. Αποχές ε, 320 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε και πάλι. Δεν ήταν σαφές. 320. Πέρασε. Εγκρίνεται. Συμβαστική 17 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. 3-2-3 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1. Και τροπολογία 324. Και θα ξέρετε τι λέει η προφορική τροπολογία Έχετε αντίληση για την ψήφιση της όχι. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 3.25 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 3.25 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 3.26 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Συμβαστική 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3.42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3.43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3.47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 3.48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3.51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 3.52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 3.49 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 3.50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3.53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3.54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3.55 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 3.59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3.60 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Επίσης συμβαστική 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 31 υπέρ. Συμβαστική υπέρ κατά αποχές συγκρίνεται. 371 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. 372 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 374 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 378 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. συμβασκή 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 386 και 387 μαζί. Είναι μας υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται. 388 υπέρ. Κατά αποχές ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά. 388. I close the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 κατά αποχές απορρίπτεται 33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 34 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται προφορική 2 και τροπολογία 41. Δεν έχετε αντίρρηση για την ψήφιση. Ψηφίσουμε υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 42 και 43 μαζί. Είναι ταυτόσιμες. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 44 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 45 υπέρ. Κατά. Αποχές εκκρίνεται. 46 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 56 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 57 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστή 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 59 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 61 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 63 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 38 συμβαστική υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 64 υπέρ, κατά υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 65 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 67 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 69 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 66 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 71 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 73 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 74 υπέρ κατά αποχές απόλυτου 75 υπέρ κατά αποχές απόλυτου 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 78 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική 39 υπέρ <clears throat> κατά αποχές εγκρίνεται 87 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 88 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 89 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 90 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 92 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 91 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 93 υπέρ κατά <coughs> αποχές εγκρίνεται 96 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 95 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 97 υπέρ κατά αποχές ε, δεκτή 94 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 98 υπέρ κατά απο αποελέγξουμε. Μία καινοτομία λοιπόν σπάσουμε τη μονατονία. 98 ηλεκτρονικός έλεγχος. Πέρας φοφορία. Απέριπτε. 99 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 100 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 101 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 102 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 103 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 104 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και η τελική ψηφοφορία στο σύνολο της έκθεσης όπως τετροποποιείται με ε, ονομαστική κλίση λέει ο πρόεδρος. Πέρας της ψηφοφορίας ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Συγχαρητήρια στους δύο συνεισηγητές για το σκληρό τους έργο. Δεν είναι εύκολο μεταξύ δύο επιτροπών να συμφωνήσουμε σε όλα τα επίμαχα σημεία και τις συμβαστικές τροπολογίες. Συγχαρητήρια στους συνεισηγητές και τις, τους σκιώδεις Έχουμε δημιουργήσει κάτι, όπως είπε και η κυρία Κώστα, έχουμε δημιουργήσει νησίδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί έτσι δουλεύει με τα κλάστες, με τις νησίδες, τα συμπλέγματα ή οι κομισιόν. Ήταν απαραίτητο λοιπόν να κάνουμε το ίδιο και μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και χαίρομαι πάρα πολύ που η συνεργασία μεταξύ των δύο επιτροπών μας ήταν επιτυχής και ήταν πολύ καλή ανταλλαγή απόψεων και οι δύο εισηγητές ήταν πραγματικά θαραλέοι και μπορούμε, μπορέσαμε να καταγάγουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ κύριε Κώστα που μπορέσαμε να επιτύχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Μεγάλη χαρά και για μένα κύριε Μπούζεκ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τα μέλη και των δύο επιτροπών για την κοινή τους προσπάθεια και να συγχαρώ τους συνεισηγητές και τους κοιόδους εισηγητές. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και τις δύο γραμματείες για την υποστήριξή τους και τις ομάδες για την έγκριση αυτή του σχεδίου εκθέσεως. Φαντάζομαι ότι οι δύο συνεισηγητές θα ήθελαν να πούν κάτι εδώ. Επίσης μετά από αυτή την ψηφοφορία, την πολύ καλή ψηφοφορία, ο κύριος Χέλλερ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λίγη ησυχία λέει κυρία Κώστα παρακαλώ. Κυρίε και κύριοι ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να τονίσω ότι δοθέντως ότι για πρώτη φορά οι δύο επιτροπές συνεργάστηκαν θεωρήσαμε ότι θα ήταν πιο περίπλοκη η διαδικασία λόγω της φύσης των επιτροπών και της συνεργασίας. Συνεργαστήκαμε ως τέλεια και ήταν κάτι εξαιρετικό και ίσως να μην είναι η τελευταία φορά που συνεργαστήκαμε διότι για πρώτη φορά καλύψαμε βρυφάσμα ε, διάφορους λόγους συλλογή δικαιωμάτων, ηθοποιούς, λογισμικό, ε, βιομηχανία παιχνιδιών, βιομηχανία, βρείτε το φάσμα. Άρα είναι η χαραυγή ενός νέου βιομηχανικού τομέα με μεγάλες προοπτικές πέρα από τις οικονομικές. Είναι ένα κομμάτι του πολιτισμού μας και ίσως ε, για πρώτη φορά ήταν ένα κομμάτι αυτό με το οποίο ασχοληθήκαμε επανέφερε και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφερόταν στην όλη κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Ένωση. Ξέρουμε ότι όλοι όσοι είμαστε εδώ έχουμε εμπειρία και θεωρούμε την έκθεση πρωτοβουλίας, πώς να το πω, ότι αναφέρει περισσότερο φιλοδοξίες παρά συγκεκριμένα πράγματα όπως νομοθεσία και χρήματα. Αλλά μάλλον το αντίθετο συμβαίνει, διότι οι διαθέταμε πραγματικά χρήματα του Ταμείου ΕΕΦΣΗ ε, για αυτόν τον τομέα και είχαμε ακόμα ασχοληθεί με αυτό το θέμα πριν ψηφιστούν αυτά τα κονδύλια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν μπορούσαμε να εκτιμήσουμε και τα αποτελέσματα της Κοινής Επιτροπής. Ευχαριστώ τον κύριο Μοργάνο, τις γραμματείες και ευχαριστώ και το γραφείο μου, την Ίνα Φερούτσι και τους ομολόγους της στο γραφείο του κ. Μοργάνο που διοργάνωσαν την όλη προσπάθεια. Δέθηκαν μεταξύ τους δύο επιτροπές, συμφωνήσαμε συμβαστικές ε, τροπολογίες και τελικά άξιζε τον κόπο αυτή η προσπάθεια και αυτή η συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θέλω να δώσω ευχαριστίες. Ευχαριστώ τον συνάδελφο Έλλερ όλους τους κοιόδης εισηγητές, τις δύο γραμματείες και πρέπει να πω και ευχαριστώ και τις δύο επιτροπές διότι έδωσαν μεγάλη προσοχή σε αυτήν την έκθεση πρωτοβουλίας. Πιστεύω ότι το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας είναι η σημαντικότερη πτυχή από πλευράς πολιτικής λόγω του τρόπου που είχε τελική ψηφοφορία και δίνει σαφές μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμπαγής μας τοποθέτηση. Δηλαδή ότι πρέπει να πρικοδοτηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση με πραγματική βιομηχανική πολιτική για την πολιτισμική και ε, δημιουργική δημοκρατία. Χρειάζεται λοιπόν μια συνεκτική πολιτική με μακροπρόθεσμους στόχους και έχουμε και χρονοδιαγράμματα όσον αφορά τα θέματα κονδυλίων του προπολογισμού και της χρηματοδοτήσεις. Είναι ένα χρονοδιάγραμμα με κοντινές ημερομηνίες και πρέπει να μπορέσουμε τελικά να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις που αμοιβαία αναλάβαμε για να ακολουθήσουμε αυτόν τον δρόμο. Θεωρώ ότι αυτό το θέμα υπησέρχεται σε μια πτυχή κοινή για όλους. Θέλουμε ανάπτυξη. Είπαμε επανειλημμένα ότι είναι από τις πραγματικές πτυχές επαναβιομηχανοποίησης της Ευρώπης που δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα, αλλά είναι πολύ σημαντικό θέμα και πίσω από αυτό πιστεύω ότι υπάρχει κοινή ένωση των προσπαθειών στο Κοινοβούλιο. Θέλουμε δηλαδή να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στην απασχόληση και κυρίως στην απασχόληση των νέων και αναφέρω πιο συγκεκριμένα και στο ότι εδώ αναφερόμαστε σε απασχόληση των νέων και στην επαγγελματική κατάρτιση και στο μέση εκπαίδευση και στην ανώτερη εκπαίδευση. Δηλαδή είναι ένα κάτι ε, που έχει στόχους μακροπρόθεσμους και ε, αυτή η προσέγγιση οδηγεί στον πραγματικό πλούτο της Ευρώπης. Ευχαριστώ όλους και εύχομαι να κάνουμε τα πάντα για να προχωρήσουμε στον τομέα. Και κλείνω λέγοντας κάτι που θεωρώ σχετικό. Έχουν εγκριθεί και άλλα πράγματα, υποστήριξη της μικρομεσαίας, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο Κοινοβούλιο και των πολύ μικρών επιχειρήσεων και τα δικαιώματα της πνευματικής ιδιοκτησίας καλύψαμε και θα πρέπει σε όλα αυτά να δώσουμε κάποια ε, προσοχή και να οδηγηθούμε σε πραγματικά αποτελέσματα. Αυτά αφορά βέβαια και άλλες επιτροπές. Ευχαριστώ λέει κύριε Κώστα. Δράτω με τις ευκαιρίες που έχω τώρα και το μικρόφωνο να πω κάτι στη μητρική μου γλώσσα. Θέλω να πω ότι ευχαριστώ τον κύριο Μπούζε και ήταν πολύ σκληρή δουλειά, δεν ήταν εύκολη διαδρομή, διότι πραγματικά έχουμε συνηθίσει σε αυτό το κοινοβούλιο, όχι μόνο στι επιτροπέ, να εργαζόμαστε κάπω απομονωμένα. Και πιστεύω ότι αυτή η προσέγγιση πιο εγκάρσια, πιο οριζόντια, χωρί βέβαια να χάνουμε τι ιδιαιτερότητε που έχει η κάθε επιτροπή. Και ευχαριστώ του ε, συγκητέ που διατήρησαν αυτή την ιδιαιτερότητα. Και η συνεργασία οδήγησε σε, ε, σε αυξημένο πλούτο για τη βιομηχανία, για το περιεχόμενο, την πνευματική διοκτησία. Επίσης και προστατεύουμε και τη μηχανή που δεν παράγει ε, τέτοια πολιτισμικά αγαθά. Λαμβάνοντας υπόψη όσες ιδιαιτερότητες, νομίζω ότι καταλήξαμε σε μια έκθεση που είναι ισχυρή. Έχουν ε, δίκιο οι δύο εισηγητές. Ε, στέλνουμε ισχυρότατο μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μέχρι τώρα Πρέπει να πω ότι ειλικρινά και μετά την πράσινη βίβλο του 2011 και την έκθεση που κάναμε προηγουμένω, δεν νομίζω ότι παρόλα αυτά μέχρι τώρα ότι έλαβε επαρκώ υπόψη ούτε στι πολιτισμικέ πολιτικέ ούτε βιομηχανικέ πολιτικέ τα χαρακτηριστικά, το DNA τη Ευρώπη που κάνει την Ευρώπη ένα αγνωρίσιμη στην Ευρώπη. Δηλαδή την ισχυρή τη δημιουργική σκέψη, του πολιτισμού, τη πολιτισμική κληρονομιά, ηλική και άλλη και των επιχειρήσεων που σε αυτό το πεδίο θέλω να υπενθυμίσω ότι υπάρχουν. Όχι μόνο βιομηχανία, και το καινού τομέα κοινωνικές επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας και αυξάνονται αυτές οι επιχειρήσεις, επεκτείνονται και δημιουργούν ποιοτική απασχόληση και συνδράμουν και στην κατάρτιση. Δεν μετακινούνται αυτές οι επιχειρήσεις, αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της κληρονομιάς και των διαφόρων περιοχών. Αυξάνεται το ενδιαφέρον για αυτές. Έχουν δημιουργηθεί σημαντικότατα δίκτυα περιφερειών που έχουν καλύψει τη δημιουργική βιομηχανία σαν ένα τομέα εξειδίκευσης που είναι συστατικό στοιχείο της εφιούς ανάπτυξης. Και στέλνουμε έτσι μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την τζιγκλίζουμε να ανταποκριθεί να κάνει κάτι όσον αφορά αυτό το τομέα στα πλαίσια του ΕΦΣΥ. Μέχρι τώρα ε, δεν έχουμε πραγματικές πλατφόρμες στο ΕΦΣΥ όσον αφορά αυτό το τομέα. Λοιπόν, αυτή θα είναι η μεγάλη μας κοινή ε, προσπάθεια και θα πρέπει να προσέξουν περισσότερο τα πνευματικά, πνευματικά δικαιώματα. Να μην θεωρηθεί το πνευματικό δικαίωμα σαν εμπόδιο στην ανάπτυξη, αλλά προπόθεση ανταγωνιστικότητα και θα έλεγα και ταυτότητα και πρωτοτυπία τη Ευρώπη στον κόσμο. Λοιπόν, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Πιστεύω ότι κάναμε μια πάρα πολύ καλή δουλειά μαζί. Υπέροχη δουλειά. Ευχαριστώ όλου, οι συγητέ, ε, του προέδρου, συμπροέδρου, ε, τι πολιτικέ ομάδε και όλου του των δύο επιτροπών, τι γραμματείε ε, που έδωσαν μεγάλη υποστήριξη. Ευχαριστώ για μια ακόμη φορά. Α, και καλώ τους συναδέλφους της Επιτροπής Πολιτισμού να εγκαταλείψουν την αίθουσα, διότι τώρα η Επιτροπή Ήτρε θα πρέπει να συνεχίσει τις δικέ της εργασίες. Ευχαριστώ πραγματικά κύριε Πρόεδρε.